μενούς εκδότες ε, στο Hong Kong. We start with the authors. First speaker, Mr. Πρώτος ο κύριος Μπουτικόφερ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Η περίπτωση των πέντε βιβλιοπολών από το Χονγκ Κόνγκ μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ειδικά καθώς έχουμε άτομα τα οποία εξαφανίζονται και μετά επανεμφανίζονται υπό μυστηριώδεις συνθήκες στην Κίνα. Και δεν μιλά μόνο για αυτούς τους πέντε. Αφορά, παραδείγματο χάρη, και έναν πρώην δημοσιογράφο της εφημερίδας Southern Metropolis Daily, τον Li Χιν και τον γιο δύο δικηγόρων ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ πως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκφράσουμε ξεκάθαρα πως αυτή η προφανώς διαδεδομένη πρακτική των απαγωγών είναι απολύτως απαράδεκτη. θα ήθελα να πω πως δύο από αυτούς τους ε, βιβλιοπόλες απολαμβάνουν τα δικαιώματα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε μας αφορά και μας. Θεωρώ πως ε, κάνουν λάθος ε, οι κινέζικες αρχές. Υπάρχει μια παλιά κινέζικη παροιμία που λέει ο βράχος τον οποίο υψώσατε θα πέσει και θα σας πλακώσει τα πόδια. Έτσι θα γίνει και τώρα. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα υποβαθμίζει το κράτος δικαίου στο Χονγκ Κόνγκ και τα επισχημένα ότι δηλαδή θα έχουμε μία χώρα και δύο συστήματα στο Χονγκ Κόνγκ και θα πρέπει η Κίνα να συμφωνήσει με τους διεθνείς κανόνες. Σας ευχαριστώ. Κοράω για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσοι μιλούν ανοιχτά και εκφράζονται ελεύθερα στην Κίνα είναι όλο και λιγότεροι ε, και όλο και λιγότεροι αυτοί που εκδίδουν. Ήδη ξεκίνησε περισσότερη λογοκρισία και καταπίεση της ελευθερίας της κοινή γνώμης ε, το 2014 και θεωρείται ότι όσοι βρίσκονται εκτός νόμου στην υπηρετική Κίνα μπορούν να καταφύγουν στο Χονγκ Κόνγκ. Όμως ε, η λαϊκή κυβέρνηση δεν ανέχεται ούτε αυτό. Ήδη η 400η ε, ε, επέτειος των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας γιορτάστηκε πρόσφατα, όμως θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση ε, η αφορμή αυτή να γίνει τρόπος να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και μόνο έτσι, με αυτή την προπόθεση, να εμβαθύνουμε τι εμπορικέ και οικονομικέ μα σχέσει. ρυθμίσει στο δικαστικό και αστυνομικό σύστημα, με τον σεβασμό τη ελεύθερη έκφραση, είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν μπορούμε να παραμένουμε αδιάφοροι, ιδίω με τέτοιε εξελίξει. Ευχαριστούμε, κύριο Παντζέρη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Του τελευταίου τέσσερι μήνε χάθηκαν τα ίχνη πέντε εκδοτών του Χονγκ εκ των οποίων ο Λίπο και ο Γκουι είναι υπηκότητας Σουηδικής και Βρετανικής. Ευρωπαίοι πολίτε απήχθησαν από τις αρχές της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας για πολιτικούς λόγους και αυτές οι εξαφανίσεις έχουν κατά πάσα πιθανότητα να κάνουν με την έκδοση λογοτεχνικών έργων που κατακρίνουν την κεντρική κυβέρνηση του Πεκίνου. Πέραν του γεγονότος ότι στην επικράτεια του Χονγκ Κόνγκ θα έπρεπε να υπάρχει ελευθερία έκφρασης, αυτή είναι μια κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι και ε, μια ε, περίπτωση μη σεβασμού των ε, πολιτικών και κοινοβουλευτικών συμφωνιών μεταξύ Κίνα και Χονγκ Κόνγκ που επιτρέπουν την ανεξαρτησία του δεύτερου κράτου. Ε, πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε και για του Ευρωπαίου πολίτε και τι άλλε προσωπικότητε, τα άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και να πάψει η αυστηρή λογοκρισία που έχει επιβληθεί με την έκδοση οποιασδήποτε επικριτική θέση στην Κίνα. Θα πρέπει η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των Κινέζικων αρχών προ τα θέματα αυτά να είναι πολύ σαφή. Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα δεχτώ γαλάζιες κάρτες γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ο κύριος Κέλαμ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τον Ιανουάριο χιλιάδες διαδήλωσαν στο Χονγκ Κόνγκ, τον Ιανουάριο τον προηγούμενο, για να εκφράσουν την ανησυχία τους ε, για την εξαφάνιση πέντε ανεξάρτητων εκδοτών και βιβλιοπολών που απήχθησαν και τους πήγαν στην υπηρετική Κίνα. Και οπωσδήποτε είναι μια ανησυχία με την οποία ε, συμφωνούμε και εμείς. Το Χονγκ Κόνγκ ε, έχει εσωτερική αυτονομία στο πλαίσιο της συμφωνίας «Μία χώρα, δύο συστήματα» που προβλέπει ελεύθερο λόγο και ελευθερίες των πολιτών. Θα θέλαμε λοιπόν να υπενθυμίσουμε στις αρχές του Hong Κόνγκ πως η ανεξαρτησία εκδοτών, blogger και βιβλιοπολών πρέπει να διασφαλιστεί και να ασχοληθούν, ε, να σταματήσουν αμέσως οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Μπέλτερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. προετοιμαζόμενος για αυτή την ε, συζήτηση στην γνωστή εφημερίδα του Hong Kong ε, South China Post ε, σε... και διάσα ένα αστείο. Το αστείο έλεγε ο καλύτερος τρόπος να διασχίσει κανείς τα σύνορα με την υπηρετική Κίνα είναι να ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο και χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα γίνεται αυτό. Δείτε πώς τα κατάφερε ο Λίμπο. Και πράγματι θα πρέπει όσοι ασκούν κριτική πλέον στο καθεστώς να προσέχουν όλο και περισσότερο. Γιατί και οι δημοσιογράφοι της South China Morning Post έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα κατάφορες παραβιάσεις της αρχής μια χώρα δυο συστήματα. Παρά τα οικονομικά μας συμφέροντα θα πρέπει να βοηθήσουμε την Κίνα σύμφωνα με την αρχή Divide and Trade. Σας ευχαριστώ. Σάντσεφ Καλτεντέι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και αδιαίρετα. Αυτό θα πει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να ισχύει για όλα ε, ανεξαιρέτως. Δεν μπορεί να σεβόμαστε μερικά δικαιώματα και άλλα όχι, ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετούμε. Εδώ δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μόνο μερικά δικαιώματα κάποιων συγκεκριμένων ε, πληθυσμών βεβαίω. Έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που επικρατούν στην Κίνα ω προ τι πολιτικέ ελευθερίε. Όμω η ελευθερία τη έκφραση θα πρέπει να ε, γίνεται σεβαστή και στην Κίνα. Το ίδιο και ο πληθυσμό των ΛΟΑΔ που ε, παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του γνωρίζουν καθημερινά. Επίσης 200.000 ε, γυναίκες ε, που έχουν μεταναστεύσει από αλλού ζουν σε συνθήκες ε, ιονής κλαβιάς ως καθαρίστριε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οικιακέ βοηθοί. Θα πρέπει λοιπόν να ένα υπερασπισμό στα του πάντε, όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριο Φαρία για ένα λεπτό. Πρόεδρε, πέντε δημοσιογράφοι και εκδότες που, που είναι γνωστοί για την έκδοση επικριτικών βιβλίων για τις κινέζικες αρχές έχουν συλληφθεί και μάλλον έχουν ε, εξαφανιστεί από το Χοκόγκ σε συνθήκες που είναι τελείως μυστηριώδες. Έχουμε μία χώρα με δύο συστήματα στο Χονγκ Κονγκ. Αυτό επιτρέπει την καταστολή βασικών ελευθεριών από τις κεντρικές κινέζικες αρχές. Ε, η περίπτωση του Xi Jinping είναι μία από τις πρώτες εκδοτών που, ε, των οποίων οι ελευθερίες καταστέλλονται στην επικράτεια του Χονγκ Κονγκ. Και κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο θα πρέπει οι αρχές ασφάλειας της Κίνας να μην μπορούν ανεξέλεγκτα να δρουν στην πρώην Βρετανική απικία του Χονγκ Κόνγκ και γι' αυτό να λάβει μέτρα και το κράτος του Χονγκ Κόνγκ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να καλέσει το Χονγκ Κόνγκ ακριβώς να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης και την άσκηση πολιτιστικών δικαιωμάτων. Το ίδιο και στα πλαίσια του ΠΟΕ και εκεί θα πρέπει να εξεταστεί και το καθεστώς ο χαρακτηρισμός της Κίνας ως αγο... οικονομίας της αγοράς. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε τους, με τους αγορητές από τις πολιτικές ομάδες και τώρα οι υπόλοιποι μιλητέ, αγορητές, ο κύριος Βέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία ε, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η Κίνα έχει προβλήματα, η οικονομική ανάπτυξη καθυστερεί στην Ταϊβάν τις εκλογές ε, την κέρδισε ένας που λέει πως πρέπει να σταματήσει η κινέζικη επιρροή στην ίσο και μετά εξαφανίζονται και πέντε εκδότες υπό μυστήριες συνθήκες. Φαίνεται πως απήχθησαν ε, γιατί ασκούσαν κριτική στις αρχές ε, του Πεκίνου. Η εξαφάνισή τους σοκάρισε το Χονγκ Κόνγκ τον Ιανουάριο. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο διαμαρτυρώμενοι κατά των απαγωγών. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέλλον της ελευθερίας ε, του Χονγκ Κόνγκ ε, και του κανόνα μια χώρα δύο συστήματα. Στο ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ζητάει από την Κίνα και το Χονγκ Κόνγκ να ερευνήσει το θέμα. Κύριε Λάινεν, ένα λεπτό. Ναι, κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με την αρχή μια χώρα δύο συστήματα και το άρθρο 27 του Basic Act το Πεκίνο έχει δεσμευτεί ε, για ελεύθερη επικοινωνία και έκφραση των ε, ανθρώπων στο Χονγκ Κονγκ. Γι' αυτό είναι ενοχλητικό να υφίστανται επιθέσεις οι άνθρωποι που γράφουν επικριτικά σχόλια. Και βεβαίως η υπόθεση αυτή είναι παγκοσμίω ανησυχητική για το εάν ισχύουν ε, ακόμα οι εγγυήσεις που είχε δώσει το Πεκίνο δεν απαγορεύεται η έκδοση βιβλίων στο Χονγκ Κόνγκ, οπότε δεν έκαναν κάτι το παράνομο αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση στο Χονγκ Κόνγκ και στο Πεκίνο να μας δώσει πληροφορίες για το πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και αν δεν έχουν κάνει τίποτα να αφαιθούν ελεύθεροι. Ζητάμε και από την Υπηρεσία εξωτερική δράση να ρίξει φω ε, στην υπόθεση και να κινητοποιηθεί για την απελευθέρωση των βιβλιοπολών. Τώρα για το KTDI θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε στο δυνατόν περισσότερους. Ξεκινάμε την κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εξαφάνιση των πέντε βιβλιοπολών από τον ίδιο εκδοτικό οίκο έχει δημιουργήσει φρίκη και τρόμο στο Χονγκ Κόνγκ. Ε, είναι επικριτικός αυτός ο εκδοτικό ε, οίκος ε, κατά του καθεστώτος στην υπηρετική Κίνα, αυτό είναι γνωστό τα βιβλία που εκδίδονται ε, είναι εχθρικά προς ε, την κυβέρνηση. Η υπόθεση Λίμπο δημιουργεί ιδιαίτερες ανησυχίες ε, διότι εξαφανίστηκε σε μυστηριώδεις συνθήκες από το σπίτι του στο Χανκ Κόγκ. Τρεις άλλοι υπάλληλοι ήταν στην Νότια Κίνα όταν εξαφανίστηκαν και αυτές οι απαγωγές είναι μια παράδεκτη πρακτική. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος για αντίθετες απόψεις. Επαραβιάζεται λοιπόν το σύστημα της μίας χώρας και των δύο συστημάτων από την Κίνα και έτσι καταπατά την ελευθερία ε, έκφρασης και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τον προηγούμενο μήνα πέντε γνωστοί εκδότες του Χονγκ Κόνγκ εξαφανίστηκαν. Ήταν γνωστοί για την κριτική που ασκούσαν στην κυβέρνηση του Πεκίνου, για τα παρασκήνια της κινεζικής εξουσίας και για διάφορα σκάνδαλα. επομένως είναι δεδομένο ότι η κοινή γνώμη του χονγκ κονγκ είναι πλέον πεπισμένη ότι υπεύθυνη για την εξαφάνιση αυτών των πέντε γνωστών εκδοτών είναι η ηγεσία του πεκίνου για τον λόγο αυτό έχουν μάλιστα και αρκετέ διαμαρτυρίε κατοίκων του χονγκ κονγκ ενάντια στην κυβέρνηση τη Κίνα, με αίτημα την απελευθέρωση των αγνοωμένων αλλά και την εμπέδωση του δικαιώματο ελευθερία έκφραση λόγου. Επομένω, η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αντιταχθεί στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνει η χώρα στο χονγκ κονγκ να υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου και τη έκφραση των εκδοτικών οίκων των δημοσιογράφων και των πολιτών τέλος όλα τα κράτη μέλη της ένωσης θα πρέπει να απαιτήσουν να εξεταστεί διεξοδικά η συγκεκριμένη εξαφάνιση των πέντε εκδοτών. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο για να υποστηρίξω την πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλαν οι συντάκτες που αναφέρατε. Ε, δύο είναι τα ζητήματα. Η τύχη των ε, πέντε ναι. βιβλιοπολών που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς ε, θα πρέπει να απιέσουμε την Κίνα ώστε να εξηγήσει ποια είναι η εμπλοκή της σε αυτή την υπόθεση και να μάθουμε τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους. Και δεύτερον, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ακριβώς τι γίνεται με τις σχέσεις υπηρετικής Κίνας και Χονγκ Κονγκ και ε, γίνεται σεβαστό το σύστημα ενός κράτους σε δύο συστημάτων, ναι ή ου. Συστηματικές παραβιάσεις ε, των δικαιωμάτων του Χονγκ από πλευράς ε, της Κίνας, καταστολή των κινημάτων για τον εκδημοκρατισμό του Kong. Αυτά τα πράγματα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Κίνα σήμερα δεν έχουν ε, εξαφανιστεί μόνο πέντε εκδότες, πέντε βιβλιοπόλες. Έχει χαθεί πλήρως και έχει παραβιαστεί τελείως, έχει κατακριμνιστεί το σύστημα των δύο χωρών, δύο συστημάτων. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, συνάδελφοι, δεν υπάρχει καθόλου. Το καθεστώς έχει ε, πλέον Ε, έχει πλέον ε, δεν έχει κανένα σεβασμό για την ελευθερία έκφρασης και η γεωπολιτική, το γεωπολιτικό βάρος της Κίνας δεν θα έπρεπε να ε, καθορίζει τη συμπεριφορά μας τα άτομα αυτά έχουν εξαφανιστεί υπό συνθήκε άγνωστε και κατά πάσα πιθανότητα ομολογίε του θα αποσπαστούν με βασανιστήρια. Πρέπει λοιπόν να καλέσουμε την Κίνα να σεβαστεί τι διεθνεί συμφωνίε που έχει συνάψει και φτάνει με τη διπρόσωπη Ευρώπη. Για μια φορά είμαστε εντελώ συνεπεί με τι αρχέ που υποτίθεται ότι προασπιζόμαστε. Ευχαριστούμε κύριο Πόλτσακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προσωπικά πιστεύω πως αυτή η βιβλιοπόλες που έχουν εξαφανιστεί είναι μία μόνο περίπτωση, ένα μόνο παράδειγμα ε, κατάφορης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα αλλά και στο Χονγκ Κονγκ. Και μετά την ε, μετάβαση στην Κίνα του Χονγκ Κονγκ βλέπουμε να προκύπτουν σοβαρά προβλήματα, διότι δεν υπάρχει πλέον όπως ε, πριν στο Hong Kong σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντίθετα καταπατούνται διαρκώς, ε, συστηματικά από την Κίνα. Και το έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένα. Θα πρέπει να απευθύνουμε και πάλι θερμές εκκλήσεις ε, για την εφαρμογή του στήχους που δέχτηκαν όταν ανέλαβαν το Χονγκ και το παρέλαβαν από το Ηνωμένο Βασίλειο ευχαριστώ. Σήμερα στο Χονγκ Κονγκ υπάρχουν παραβιάσεις των συνταγματικών κανόνων, συλλήψεις, εξαφανίσεις ε, βιβλιοπολών και εκδοτών που ε, λόγω αυτών που εκδίδουν και μεταπολούν, χρησιμοποιούν προσχήματα όπως ε, οδήγηση σε κατάσταση μέθης, παραδείγματος χάρη και τελικά εξαφανίζουν σε παράνομους χρόνους κράτησης. Ε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ε, πλέον επίσημα ότι το καθεστώς, δηλαδή μία χώρα, δύο συστήματα, παραβιάζεται από πλευράς της Κίνας και υφίστανται διακριτική μεταχείριση ε, οι κάτοικοι του Χονγκόγκα και γι' αυτό θα πρέπει να τους ε, βοηθήσουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το διπλωματικό εργαλείο που έχουμε στις σχέσεις μας ε, με την Κίνα, ούτω ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνω τη διαδικασία Κατσίαη και τώρα η κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Εξακολουθούμε να μην έχουμε ακριβείς πληροφορίες ε, για την κατάσταση αυτών των βιβλιοπολών ε, που συνδέονται με τον εκθετικό οίκο με την ε, και ανησυχούμε ιδιαίτερως. Γιούμιναϊ ε, από το Σουδάν, ε, Λίποι ε, από τη Βρετανία είναι και σε ειδικότητα, δηλαδή κάποιοι από αυτού, και από τη αμέσα Οκτωβρίου έχουν να ειδωθούν οι δύο από αυτού στην Ταϊλάνδη. Παραβιάζεται το Σύνταγμα αν οι αρχές επιβολής ε, του νόμου όντως ε, της υπηρετικής Κίνας έχουν δράσει κατά αυτόν τον τρόπο στο Χονγκ Κονγκ. Ε, μία χώρα, δύο συστήματα, αυτή είναι η αρχή που πρέπει να γίνεται σεβαστή, όμως δεν γίνεται και είναι ελεύθερη η κοινωνία και θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία έκφρασης στο Χονγκ Κονγκ, στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη. Θα πρέπει ανεξάρτητες αρχές να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εξαφανίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι βάσει των αρχών του κράτους δικαίου. Είπα ότι εκπρόσωπος ο Μογκερίνη έκανε σχετική δήλωση για την εξαφάνιση ε, των όσων συνδέονται με τον εκδοτικό εκομμάτι κάνω στο Χονγκ Κόνγκ τον Ιανουάριο. Είμαστε σε επαφή με τις αρχές του Χονγκ Κόνγκ και συνεργαζόμαστε στενά και με το Ηνωμένο Βασίλειο τη Σουηδία επίσης ε, και τους επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Χονγκ Κόνγκ για αυτό το ζήτημα. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από το Πεκίνο πληροφορίε από τις ε, κινέζικες αρχές. Προς το παρόν ε, δεν έχουμε αξιόπιστες ε, ακριβείς πληροφορίες παρότι τις ζητήσαμε και το ίδιο σημαίνει και με την αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου επί τόπου. Θέλουμε να διευκρινίσουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται όσοι συνδέονται με τον εκδοτικό οίκο ε, Mighty και θα πρέπει να δοθεί πρόσβαση στις προξενικές αρχές για τους ξένους επικόρους που έχουν εξαφανιστεί. Ε, ευχαριστώ. Έχω, θα εγκρίνουμε μετά τη συζήτηση